Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 5ης Φεβρουαρίου έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσει σχετικά? Ο Τζάζ Τσίσεστερ, παρακαλώ. Uh, um, Κύριε Πρόεδρε, όχι για τα πρακτικά, αλλά σαν πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία είπατε και θα μεταφέρουμε το μήνυμά σας την επομένη εβδομάδα στην Αυστραλία. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν επόμενε παρατηρήσει σε σχέση με τα πρακτικά. Θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Στι 9 Δεκεμβρίου 2008, ο κύριο Βίτολ Τόμτσακ έχει κάνει μια αίτηση για την διατήρηση